Présidente. Bien, merci, chers collègues. Nous allons. Euh, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Κόμι έχεις δει το λόγο. Αλλά παρακαλώ καθίστε για να ακούσουμε την κυρία Κόμι. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Κόμη. 186 Αναφέρομαι στο 186 του κανονισμού. Μετά από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ινδίας που απέρριψε ε, την έφεση των δύο ναυτικών ε, Ιταλών που για λόγους υγείας πρέπει να παραμείνουν στην Ιταλία. Ε, έχουν παρέμβει στο παρελθόν οι Άστον και άλλοι, ζητάμε από τη Μογκερίνη το ίδιο. Οι πολίτες αυτοί, οι δύο αυτοί ναυτικοί είναι συμπολίτες μας, πρέπει να τους φροντίσουμε. Euh, Κύριε Μπασίρ, 30 δευτερόλεπτα. Διαδικαστικό. Συνειδητοποιείτε ότι έγινε, συνέβη μια τραγωδία στο Πακιστάν, στο Πεσαβάρ. 500 άτομα αυτή τη στιγμή είναι όμοιροι. 124 παιδιά σκοτώθηκαν, 200 παιδιά είναι τραυματίες. Αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τους ε, ακραίους, τους εξτρεμιστές, όχι για να προστατεύσουμε το Πακιστάν, αλλά για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Πρέπει να αποστείλουμε ένα μήνυμα συμπάθειας και κατανόησης ε, σε αυτό τον λαό για να βρει τη δύναμη να καταπολεμήσει την απειλή των Ταλιμπάν. Πρέπει λοιπόν όλοι χωρίς εξαιρέσεις να βοηθήσουμε τη χώρα να καταπολεμήσει τους εξτρεμιστές. Σπινέλη, τελευταίο διαδικαστικό πριν ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Εξ ονόματος των Ιταλών μελών της ομάδας Γκουε θα ήθελα να σημειώσω κάτι το πάρα πολύ σοβαρό που συνέβη στις 15 Δεκεμβρίου. Ένας γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος τελευταίος μέλος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Κέζα, συνελήφθη στο Ταλίν στην Εσθονία πριν πάει σε μια δημόσια συνάντηση στην οποία είχε προσκληθεί. Ελευθερώθηκε, εκδόθηκε στην Ιταλία ε, ως μη επιθυμητό πλέον πρόσωπο στην ε, συγκεκριμένη χώρα. Ε, τίτλος της συνάντησης αυτής την οποία πήγαινε ο κύριος Κέζα ήταν «Η Ρωσία ο εχθρός μας» με ερωτηματικό. Λοιπόν, σε μια ευρωπαϊκή χώρα απαγορεύθηκε να πάρει τον λόγο δημόσια. Δεν ήταν και πολύ διαδικαστικό λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο θέμα της εκλογής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Σύμφωνα με το 219 Έχω την υποψηφιότητα της κυρίας Έμιλι Ορέιλι. Σύμφωνα με το άρθρο 219 παράγραφος 5 η ψηφοφορία θα είναι μυστική και πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία των εκπεφρασμένων ψήφων και οι αποχές δεν θεωρούνται τέτοιες. Λοιπόν, πρόκειται για μυστική ψηφοφορία. Αυτό σημαίνει ότι θα ανάξει το μπλε φωτάκι στην κονσόλα σας ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσετε. Σύμφωνα τώρα στην παράγραφο 6 του 2019 πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τα μισά μέλη του Κοινοβουλίου. Βέβαια αυτό ισχύει και γι' αυτό θα, υπάρξουμε, θα υπάρξει δοκιμαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, δοκιμαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Τεστ κύριε, μη διαμαρτύρεστε, τεστ Λοιπόν, ε, είναι επαρκής ο αριθμός, υπάρχει απαρτία και περνάμε τώρα στην εκλογή της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Σας έχετε το λόγο. Ε, μπροστά από μένα υπάρχουν δύο μηχανές οι οποίες ε, δεν δουλεύουν, δύο κονσόλες που δεν δουλεύουν. Πρέπει να έρθει ένας τεχνικός. Ναι, θα σας το επισκευάσουμε λέει η Πρόεδρος. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία τώρα για την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Tout le monde a-t-il voté? Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 569 suffrages positifs. 569 υπέρ, 66 κατά, 43 αποχές. Euh, euh, euh, λοιπόν, η πλειοψηφία τίμησε την κυρία O'Reilly. Είναι διακηρύσω πλέον Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια. Σύμφωνα με το άρθρο 7, το άρθρο 219, παράγραφος 7. Συγχαρητήρια κυρία Ρέιλι. Περνάμε τώρα τις ψηφοφορίες των εκθέσεων. Πρώτη είναι η έκθεση του κυρίου Λαβία, επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Συγχαρητήρια κύριε Λαβία. Σύσταση της κυρίας Σαγιούζο για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, ΣΥΤΕΣ. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας, δεκτή. Περνάμε τώρα στην σύσταση Μπούζεκ για τη Συμφωνία Συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα με το Μαρόκο. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία. Περνάμε τώρα στη σύσταση Μπούζεκ για την ανανέωση της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με την Ουκρανία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. Δεκτή. Περνάμε τώρα στη σύσταση Λάμστορφ για τη συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μία η ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή η πρόταση Λάμστορφ. Έκθεση της κυρίας Μιχαήλοβα για την εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές απόκεντρες περιοχές. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραστη της ψηφοφορίας. Δεκτή η πρόταση. Περνάμε στην έκθεση βιώτη για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής. Εδώ απαιτείται ειδική πλειοψηφία των τριών πέμπτων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραστη της ψηφοφορίας. Δεκτή η πρόταση. Έκθεση Όλμπρεκ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Fiat Πολωνίας. Ονομαστική ψηφοφορία, ειδική πλειοψηφία τριών πέμπτων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Περνάμε τώρα με την έκθεση Βάναμ κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου σχετικά με την Οδυσσεύς Φωκάς. Τρία πέμπτα απαιτούνται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή η πρόταση Βάνα. Περνάμε τώρα στην έκθεση Τζάνι πάντα για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση σχετικά με την Εμφρόνς. Απαιτείται πλειοψηφία τριών πέμπτων. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή και η πρόταση Ζάνη. Τελειώνουμε με την έκθεση Γκουαλτιέρη σχετικά με το διορισμό μέλους του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Τραπεζών. Μία ψηφοφορία, νηστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Le vote est clos. Πέρα και η συγκεκριμένη έκθεση γίνεται δεκτή. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. D'accord.